Okay, dear colleagues, we have rapporteur and then... Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε έναν εισηγητή και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ε, πρώτο σημείο είναι η έγκριση της ημερήσιας διατάξεως. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνουμε χωρίς αλλαγές την ε, ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις του Προέδρου, σημείο 2. Έχουμε ένα διορθωτικό στην οδηγία 40-2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2013 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σε σχέση με την ε, μεταποίηση και πώληση καπνού και προϊόντων καπνού ε, ήταν μια οδηγία που τροποποιούσε την 37 του 2001. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησε θέση στον πρώτη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου. Το σφάλμα αφορά μια ε, ε, λάθος αμνία στο σημείο F, σημείο δε, ε, ε, παράγραφος 10. Το διορθωτικό εστάλει σήμερα το πρωί. Αν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται αυτό το διορθωτικό και θα το υποβάλουμε στην, στο Κοινοβούλιο ώστε να ανακοινωθεί στη δεύτερη σύνοδο του Απριλίου. Δεύτερη ανακοίνωση, εργαστήριο για τους δείκτες ε, επάρκειας πόρων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας της κυρίας Φιετικάινεν που αφορά την ε, επάρκεια των πόρων. Αυτό θα γίνει αύριο στις 14 Απριλίου στις 12.30 12.45 ε, συγγνώμη, στην αίθουσα ASP 1Ε2. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ε, Πολιτών για, την, για τα πειράματα σε ζώα υπευλήθη ε, η Επιτροπή ε, Γεωργίας θα διοργανώσει σχετική ακρόαση, η ΕΜΒΙΤΡΙ και η ΠΕΤΗ θα συνδεθούν και η ακρόαση θα γίνει στις 11 Μαΐου 2015 στην αίθουσα 4 και 2. Σχέδιο προγράμματος και σχετικές πρακτικές ρυθμίσεις θα κυκλοφορήσουν ε, συντόμως. Σήμερα έχουμε διερμηνία σε 22 γλώσσες, δηλαδή λείπουν τα εστονικά και αύριο θα έχουμε διερμηνία σε 21 γλώσσε. Όσοι ήθιστε, η συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 3ης και 4ης Δεκεμβρίου και της 21ης και 22ης Ιανουαρίου. Είναι έτοιμα τα πρακτικά. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται αυτά τα πρακτικά. Σημείο 4. Θα πρέπει να σας ενημερώσω σχετικά με τις συνεχιζόμενες διοργανικές διαπραγματεύσεις. Έχουμε τον πρώτο άτυπο τριμερή διάλογο για το σύστημα ITS, σχετικά δηλαδή με το σύστημα σταθερότητας ε, για την, της αγοράς ε, έγινε στις 23 Μαρτίου. Κάναμε μια ε, σοβαρή ανταλλαγή απόψεων για τα πολιτικά θέματα που διακυβεύονται. Παρά την σημαντική διάσταση απόψεων, η συζήτηση έγινε σε επικοδομητικό πνεύμα και συμφωνήθηκε να αναθεθούν στο τεχνικό επίπεδο για περαιτέρω εξέταση κάποια ζητήματα πριν από το δεύτερο τριμερή διάλογο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα εξή θέματα. Ε, έναρξη του αποθεματικού σταθερότητας αγοράς, η ε, ποσοστώσεις, ε, οι προκαταβολικές ποσοστώσεις, το Ταμείο Καινοτομίας και η διαρροή άνθρακα. Η δεύτερη στιγμερή θα γίνει στις 5 Μαΐου, στις 4 η ώρα. Τώρα πάμε στο σημείο 5. Μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρήπων και τροποποίηση της οδηγίας. Έχουμε τον εισηγητή μας, την εισηγήτριά μας εδώ και θα ξεκινήσουμε αμέσως. Σας δίνω το λόγο, κυρία Γκέρλιγκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα πω πολλά εισαγωγικά. Όλοι γνωρίζουμε τις στατιστικές, ποια είναι τα σημερινά ζητήματα υγείας που αντιμετωπίζουμε. Για παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν σοβαρά ζητήματα ύπασης της ατμόσφαιρας σε διάφορα σημεία της Ευρώπης. Με την σκόνη από τη Σαχάρα για παράδειγμα και η υψηλά επίπεδα ρήπανσης, κάτι το οποίο θα έχουμε αρκετά συχνά στο μέλλον αν δεν κάνουμε κάτι για να το αντιμετωπίσουμε. Οπότε, εντάξει, εγώ δεν θα αναφερθώ σε αυτό επί μακρό. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι καλά εδώ στην Επιτροπή μας. Αυτό όμως που θέλω να κάνω είναι πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την έκθεσή της και για τη δουλειά που έχει κάνει. Είναι κάτι που περιμέναμε εδώ και καιρό. Δεν είναι και κακό βέβαια αυτό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω εγώ και έχοντας συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια επί του θέματος. Έχει γίνει πολλή δουλειά για το πρωτόκολλο του Γκέτεμπορκ. Έχουν ε, δει και άλλους δείκτες, όπως τις προδιαγραφές που βάζει ε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κλπ. κλπ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχει και η απειλή της Επιτροπής που ήταν να αποσύρει την εκθεσή της, κάτι το οποίο δεν έκανε ποτέ, ευτυχώς, και έτσι συνεχίσαμε. Και σήμερα πια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς εδώ στην Επιτροπή μας μπορούμε να ε, ψηφίσουμε πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε καλό είναι που προχώρησε το θέμα. Πολύ σημαντικό γιατί είναι θέμα δημόσιο. Είναι κάτι που μας αφορά όλους όχι μόνο επειδή είμαστε μέλη της Επιτροπής αυτής, οπότε μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, αλλά και πολιτικά σε πάρα πολλές χώρες μέλη έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις στο θέμα του περιβάλλοντος και είναι ψηλά ψηλά στην ημερήσια διάταξη τα τελευταία χρόνια. Καλό είναι λοιπόν που μπορούμε να προχωρήσουμε. Πολύ καιρό έχουμε επικεντρωθεί στις εκπομπές και στα αέρια του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει γίνει χωρίς να ασχοληθούμε εξίσου πολύ και με τους ρηπαντές. Έχουμε λοιπόν πια αυτή την ευκαιρία. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω εγώ το θέμα πριν ακούσουμε τους σκιώδεις εισηγητές. Όπως σας είπα, έχω περάσει πολύ καιρό εξετάζοντας την πρόταση και τις λεπτομέρειες. Μερικές από αυτές είναι πάρα πολύ τεχνικές. Όσοι έχετε κοιτάξει τα παρευθύματα το ξέρετε αυτό. Δύσκολο τεχνικά. Είδα λοιπόν και τα παραστήματα που αναφέρουν τις ανώτατες τιμές, αλλά δεν είναι εδώ που θέλω να αναμειχθώ. Δεν είναι ότι θέλω να αλλάξω τα ποσοστά προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με τους δείκτες, τους λιπαντές κτλ. Όχι, αλλά γνωρίζουμε ότι οι χώρες μέλη συζητούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα στοιχεία αυτά. Έχουμε φτάσει σε κάποιο σημείο που υπάρχει συμφωνία επ' αυτών. Δεν θέλω λοιπόν την συμφωνία αυτή εγώ να την χαλάσω. Όμως υπάρχει κάτι στα παραρτήματα που πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Είναι η δεσμευτική στόχη για το 2020. Διαβάζοντας το μερικές φορές θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήδη είναι δεσμευτική στόχη, αλλά δεν πρέπει να μείνει καμία αμφιβολία, οπότε νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λέμε για το 2025. <clears throat> Συγγνώμη, ότι είναι δεσμευτική η στόχη αυτή. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μου θέμα. Το 2025 είναι μια σημαντική ημερομηνία, γιατί αν το αφήσουμε για το 30, είναι πολύ μακριά. Και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε, παρά τις καλύτερες προθέσεις που βέβαια έχει Επιτροπή και όλοι οι υπόλοιποι, τα κράτη-μέλη δεν θα το κάνουν. Θα πούν ότι θα το κάνουν μόνο το 2020-2025, αλλά τότε δεν θα προλαβαίνουμε. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό η συζήτηση αυτή να γίνει πριν το 2025. Είχα κι εγώ πολλές αντιδράσεις σχετικά με το δεσμευτικό αυτό στόχο του 2025. Πρέπει όμως να το κρατήσουμε νομίζω. Στην πρότασή μου Ευελτιώνω νομίζω κάπως το θέμα της ε, αναφοράς, της ενημέρωσης και της ε, ανείχνευσης. Πιστεύω ότι η πρόταση είναι καλή. Επιδέχεται βέβαια βελτιώσεις. Ένα πολιτικό ζήτημα όμως θέλω να αναφέρω. Όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολος θα αποδειχθεί ο φάκελος αυτός προκειμένου να περάσει από τη διαδικασία συναπόφασης. Και ποτέ βέβαια εγώ δεν σκέφτηκα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει να πάρει μια ακραία θέση γνωρίζοντας ότι τα κράτη-μέλη θα πάρουν μια άλλη ακραία θέση και ότι θα είναι δύσκολο να βρεθούμε ε, στη μέση και να βρούμε ένα συμβασμό. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το ποιοι είναι οι στόχοι μας και οι φιλοδοξίες μας. Πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι πάντα σε ένα βαθμό υπάρχει και η ιδέα της απόσυρσης, ότι μπορεί δηλαδή να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο της απόσυρσης της πρότασης. Να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Συνεπώς, ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να πιέσουμε τις χώρες μέλη για κάτι πιο φιλόδοξο από αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να πάμε πολύ μακριά. Να σας αναφερθώ λίγο και σε άλλη νομοθεσία και το λέω αυτό κυρίως εξαιτία τη έκθεση αντικτύπου την οποία ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι δίνει μια σαφή κατεύθυνση για τη συνέπεια που θέλουμε να υπάρχει και τη συνοχή με το πακέτο για το κλίμα. Νομίζω ότι όντω πρέπει να προσπαθήσουμε κάπως πιο γρήγορα να πετυχαίνουμε αποτελέσματα. Συμφωνώ, μεν, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι επρόκειτο για μια έκθεση αντικτύπου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δεν αξιολογήθηκε από την Επιτροπή και θα ήθελα να γίνει αυτό πριν το συμπεριλάβουμε στην νομοθεσία. Αυτή η διαδικασία όσον αφορά το πακέτο για την κλιματική αλλαγή παραμένει, συνεχίζεται. Λοιπόν, τα νούμερα είπα, δεν τα αλλάζω. Μιλάω για ένα μεκανονισμό που θα πρέπει να μας βοηθάει να ε, αξιολογούμε σε κάποιο μετέπειτα στάδιο τα νούμερα. Νομίζω ότι είναι πιο ρεαλιστικό αυτό. Ένα σημαντικό ζήτημα εδώ έχει να κάνει με την καλύτερη χρήση των πόρων. Πρόκειται για την οδηγία οροφή, η οποία έχει να κάνει με την νομοθεσία που πρέπει να είναι αποτελεσματική ώστε οι χώρες μέλη να κάνουν ε, τα δικά τους τα σχέδια αλλά να μπορούν να έχουν και κάποια βεβαιότητα. Το βασικό εδώ είναι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και το ΚΑΡΣ. Προς το παρόν, ενώ μας έχουν γίνει προτάσεις για τα θέματα αυτά και για τον ντίζελ. Εγώ ρητά στην έκθεσή μου λέω ότι πρέπει να υπάρξει κάτι γι' αυτό. Και μιλάω και για πραγματικές δοκιμές κάθε φορά που ένα όχημα αρχίζει να κυκλοφορεί. είναι κάτι που για μένα είναι σημαντικό. Ως εισηγήτρια πάντως για αυτό το θέμα, για πρώτη φορά νομίζω ως Ευρωβουλευτής πρέπει να ξέρετε ότι είχα φοβερό λόμπινγκ και από πολίτες και από περιφέρειες. Όχι μόνο από τις κυβερνήσεις των χωρών μελών που επίσης, αλλά περιφέρειες, δήμοι. Και ήταν φοβερό γιατί δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον για αυτή την νομοθεσία, γιατί αυτοί θα πρέπει να τη θέσουν σε εφαρμογή, ιδιαίτερα σε πόλεις που υποφέρουν από κυκλοφοριακή συμφόρεση και έχουν προβλήματα με την ποιότητα του αέρα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά τις δοκιμές επί των οχημάτων. Πώς να το πω, δεν θα έλεγα ακριβώς ότι είναι απελπισμένοι, αλλά ίσως αυτή είναι η καταλληλότερη λέξη. Αναρωτιόνται πώς θα το πετύχουν αυτό. Κάνω λοιπόν προτάσεις εδώ για το πώς θα έπρεπε να γίνει αυτό. Σίγουρα και άλλοι θα μιλήσουν για αυτά τα ζητήματα. Πάντως οι χώρες μέλη πρέπει να έχουν ε, τα εργαλεία στη διαθεσή τους για να κάνουν αυτή την καλή δουλειά. Τώρα, όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Όσον αφορά την αμμονία και τη γεωργία, είναι μια ρηπογόνος ουσία που εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να αποκλείσουμε από τους υποχρεωτικούς στόχους του 2025. Και θα σας πω γιατί. Δεδομένης της νέας ε, κοινή γεωργικής πολιτικής, πολλοί από εμά έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτά, εσείς ε, και η Γερμανία, και ξέρουμε πόσο χρόνο μας πήρε Ξέρω ότι υπάρχουν ε, πολλά πράγματα που ζητάνε από πλευράς ε, γερικών επιχειρήσεων για το πώς να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Θέλω να πω ότι προσθέτοντας εδώ την απέτηση αυτή για την αμμονία, που εντάξει είναι αναγκαίο, απαραίτητο, δεν το αμφισβητώ, αλλά το βάλουμε και αυτό σαν απέτηση, χωρίς να σκεφτούμε πώς θα γίνει η χρηματοδότηση γι' αυτό, θα ήταν άδικο και μη ρεαλιστικό. Τι πρότεινα λοιπόν τελικά. Πρότεινα να αποτελέσει μέρος του πακέτου στα μέσα του δρόμου του για το 2017 λοιπόν και εκεί να δούμε πού θα μπει στον κατάλογο των απαιτήσεων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις χωρίς όμως να έχουμε λύση για τη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να γίνει. Το γεωργικό λόμπι είναι πολύ δραστήριο. Τα λέει με το όνομά του τα πράγματα. Λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε. Λένε ότι δεν πρόκειται να σας βοηθήσουμε. Και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο στην Επιτροπή μας. Να φροντίσουμε δηλαδή η γεωργική μας πολιτική να είναι τέτοια που να μπορεί να λειτουργήσει μαζί με τις άλλες πολιτικές μας. Γι' αυτό λοιπόν το 2017 θα πρέπει να δώσουμε καλή κατεύθυνση από αυτού. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά πρέπει για να βγούμε από τα διέξοδο. Έχω και κάτι για την πρόσβαση στην ενημέρωση. Οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν. Οι πολίτες μας γράφουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την ρήπαση της ατμόσφαιρας τις τελευταίες εβδομάδε, για παράδειγμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Να τους δώσουμε λοιπόν ένα ρόλο να παίξουν κι αυτοί είναι σαφές ότι πρέπει να διασφαλίσουμε πως οι χώρες μέλη σχεδιάζουν αφού προηγουμένως έχουν διαβούλευση με τις διάφορες ομάδες συμφερόντων. Επίσης έχω και κάποιες ρήτρε εδώ που λέω ότι αν η νομοθεσία δεν λειτουργεί να μπορούν οι πολίτες να έχουν λόγο. Και πιστεύω ειλικρινά ότι βελτιώνοντας την συνειδητοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών, αυτό μπορεί να βοηθήσει να καταλήξουμε ε, ώστε τα μέτρα τα οποία θα επιβάλλουμε να γίνουν πιο εύκολα αποδεκτά από τους πολίτες. Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε ένα ζήτημα για το οποίο μέλη της Επιτροπής μας μου μίλησαν. Και αυτή είναι η ευελιξία shipping flexibility. Κυρίως γιατί δεν είναι κάτι που αφορά όλες τις χώρες μέλη εξορισμού. Δεν έχει να κάνει με όλες τις χώρες. Δεν θα ήταν δίκαιο λοιπόν. Πολλά λοιπόν πρόκειται για τις θαλάσσιες εκπομπές ευελιξία όσον αφορά τι θαλάσσιε ε, εκπομπές. Αλλά τότε η ευελιξία δεν θα εφαρμοζόταν ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη-μέλη, δεδομένου ότι θα αποκλείονταν οι χώρε που δεν βρέχονται από θάλασσα. Τέλο, θέλω να ευχαριστήσω του σκιώδει εισηγητέ για την βοήθειά του μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στο Better Λίζε από πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα αγγλικά και στα γερμανικά. Ευχαριστώ και την κυρία Γκέλινγκ. Ο κύριο Κίζεκερ είναι δικό μα και όδη Δυστυχώ ε, έχει κολλήσει ένα ποτηλιάρισμα. Γι' αυτό αναλαμβάνω εγώ. Ευχαριστούμε την Τζούλη Γκέρλινγκ για το σχέδιο τη έκθεσή τη και για την καλή φυσικά συνεργασία που είχαμε. Τώρα, μετά από μερικές αναταράξεις και κραδασμούς, έχουμε αρχίσει την νομοθετική διαδικασία. Είμαστε στην αρχή. Ε, δίστανται και απέχουν πολλοί απόψει και στο εσωτερικό του Έλκα ακόμα δεν έχουμε εξαντλήσει τη συζήτηση. Είναι μια πρώτη μόνο εκτίμηση του Γιάννη και του σκιώδη συγκητή μα, που θα σα παρουσιάσω ουσιαστικά προτείνει να υποστηρίξουμε την Τζούδι Γκέρλινγκ και ιδιαίτερα το πολύ ε, επίμαχο και αφιλεγόμενο θέμα της αμμονίας που το συζητάμε σφόδρα και με τους συναδέλφους της Επιτροπής Γεωργίας και προβληματίζεται ε, ο σκιώδης Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερη ευελιξία πάντα βασιζόμενη στην αρχή της επικουρικότητας και σκεπτόμενη τις ε, εξαιρέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω. Και επιπλέον η διαρθρωτική μεταρρύθμιση στην ε, η Γεωργία κινδυνεύει να διακυβευτεί από αυτή τη ρύθμιση. Καλωσορίζει την υποστήριξη, την οικονομική των αγροτών για να μειώσουν ε, τις εκπομπές και να πετύχουν αυτούς τους στόχους και παραπέμπει στο εξή γεγονό για την αμμονία πάντα να μην έχουμε διπλές ρυθμίσει. Τώρα σε ό,τι αφορά τους ενδιάμεσους στόχους για το 2025 ο κύριος Γκίζεκε θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να είναι αυτή η δεσμευτική η ενδιάμεση στόχη για το 2025. Οι στόχοι της μείωσης τώρα για το μεθάνιο είναι κάτι που το βλέπει με μεγάλη επιφύλεξη. Να μην έχουμε διπλές ε, ρυθμίσεις και με τα κλιματικά και με τα όσα συζητούμε τώρα. Αυτό που υποστηρίζει πλήρως είναι ε, η ε, διαγραφή της πρόταση για τις θαλάσσιες μεταφορές, όπως είπε και η Judy Gerling, και το θέμα του γύρω 6 για τα αυτοκίνητα. Μια που έχω το λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκέρλι για τον αγώνα που έδωσε τους τελευταίους μήνες. Ήταν πραγματικά δύσκολη υπόθεση ε, για να διατηρηθεί στη ζωή αυτή η νομοθεσία ε, και η ίδια εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά και με επιτυχία και αυτό που έχει σημασία είναι να δώσουμε συνέχεια και να διαφυλάξουμε τα όσα επιτύχαμε στην επόμενη διαδικασία και να είμαστε ρεαλιστές δεν ε, εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο της απόσυρσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τις λεπτομέρειες θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε αρκετό χρόνο και πολλές ευκαιρίες στους επόμενους μήνες. Ε, προσωπικά ε, θεωρώ πολύ πιο λογική αυτή την τακτική που ακολουθούμε τώρα, να παραμένουμε στο κείμενο, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα για να τα λύσουμε, αντί να αποσυρθεί η πρόταση γιατί υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις. Είμαστε σε καλό δρόμο με την πρόταση της κυρίας Σκιόλινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Στάντ. Κύριε Ντάνς, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ατμοσφαιρική ρήπανση στις Βεξέλλες πιάνει βήχας. Λοιπόν, θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με τον Πίτερ και να ε, συγχαρώ και εγώ την ε, κυρία Γκέρλινγκ για το έργο της. Αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο και το γνωρίζω. Παρόλο που είμαι νέος βουλευτής, <laughs> άκουσα ότι δεν είναι φυσιολογική η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα και χαίρομαι που ε, κατέληξε έτσι. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε, αλλά δεν θα την είχαμε εάν δεν ε, είχε ακολουθήσει αυτή η στάση η κυρία Γκέρλινγκ. Θα είχε αφαιρεθεί ε, το θέμα από το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ευχαριστώ και την ευγνωμονώ γι' αυτό. Επίσης την ευγνωμονώ για κάτι άλλο, για το περιεχόμενο της έκθεσης, αυτό καθ' αυτό. Θα ήθελα γενικά να σας δώσω την αίσθηση είναι μια πολύ καλή αφετηρία για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, όχι μόνο εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά και με το Συμβούλιο. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ε, ορισμένα που μας χαροποιούν πολύ. Το πρώτο είναι δεσμευτική στόχη για το 2025, είναι πάρα πολύ σημαντικό ως ε, τροπολογία. Το έχουμε συζητήσει αυτό επί μακρόν και ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους κινδύνους. Τα κράτη-μέλη να βρεθούν σε μια κατάσταση που να υποχρεωθούν να, να λάβουν δραστικά μέτρα μέχρι το 2020. Οτιδήποτε οδηγεί σε πιο ομαλή μείωση είναι πρόσδεκτο, καλοδεχούμενο. Προφανώς ε, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι κάτι που πιέζει και όσο πιο γρήγορα το λύσουμε τόσο καλύτερα για όλους γιατί μας αφορά άμεσα εδώ και τώρα. Το άρθρο 6 θέλω να παραπέμψω που ε, ενισχύει τα εθνικά προγράμματα για τον έλεγχο της ρήπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το συνδέει και με την ε, σύμβαση του Άρχους και με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και συμφωνώ με την κυρία Γκέρλινγκ. Χρειάζεται να το δούμε σωστά και να κωδικοποιηθεί στην ίδια την οδηγία. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω την αύξηση της συνοχής ε, για το πώς συνδυάζονται οι διάφορες νομοθεσίες, το ε, Euro 6 που ακούσαμε μόλις τώρα και τις εθνικές προσπάθειες για τον έλεγχο της ρήπασης του ατμοσφαιρικού αέρα. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των εκπομπών ρήπων στην πηγή τους, έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Και ο λόγος που δεν αποσύρθηκε τελικά αυτό το πακέτο, αυτή η δέσμηση, είναι ότι υπάρχει μεγάλος χώρος να συνδεθεί με άλλα νομοθετήματα στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έχουμε απόλυτο καθαρό και σαφές. Και είναι πολύ μεγάλη πρόοδος αν σκεφτεί κανείς τη σημερινή συνοχή μεταξύ. Τώρα σε ό,τι φορά τις αλάσσιες εκπομπές και την ε, αντίστοιχη ευελιξία χαιρόμαστε και υποστηρίζουμε τη διαγραφή αυτής της ρύθμισης. Ήταν περίπλοκο γιατί δεν αφορούσε όλα τα κράτη-μέλη και όπως γνωρίζουμε Είχαμε ένα επεισόδιο αυτή την εβδομάδα, ρήπανση στα, σωματίδια για τα οποία μιλούμε. Πηγαίνουν στην ατμόσφαιρα και ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα. Οπότε δεν έχει νόημα να στιγματίζεται ένας ε, τομέας, ε, ένας κλάδος οικονομίας σε σχέση με άλλους. Ε, είμαστε υπέρ αυτής της γραφής στην θαλάσσια ρήπανση. Για την αμμονία τώρα. Εδώ υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις σε σχέση με τα όσα λέει ο Πέτερ Λίζε. Η εξαίρεση λέει από τους στόχους του 25. Κατανοώ τη λογική και τις ανησυχίες που ακούγονται, ειδικά από ορισμένου ε, γεωργούς. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο που το συνδέει με την αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής το 2017. Θα πρέπει να τονίσουμε και να το τονίσουμε συνέχεια ότι φυσικά οι πόλεις ενδιαφέρονται πάρα πολύ γιατί τους αφορά το πρόβλημα Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι η κυκλοφορία στις πόλεις που αυξάνεται και ιδιαίτερα τα αυτοκίνητα diesel είναι πρόβλημα. Αλλά η αμμονία ε, είναι ένας φορέας που μεταφέρει αρουμένα σωματίδια στην ατμόσφαιρα και αυτό ε, δημιουργεί προβλήματα με τον έφος όπως έχουμε δει πρόσφατα και στο Ρονδίνο, ε, το οποίο όμως ε, νέφος μεταφέρεται και στη Βόρεια Γαλλία και με ακολουθεί και εμένα από το τρένο το Eurostar μέχρι τις Βρυξέλλες και πάει λέγοντας. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι συνδέονται αυτά τα ζητήματα, το μεθάνιο, η αμμονία και άλλοι ρηπαντές. Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τη σημασία της δράσης αυτοκού, όσο λέγει ο Πέτερ Λίζε για τις διπλές μετρήσεις, εγγραφές, αλλά το πνεύμα της οδηγίας είναι να μειωθούν συνολικά οι ρηπαντές και μέχρι το 2030. Αν συνδυαστούν οι προσπάθειες αυτές θα είναι και αποτελεσματικό, θα κερδίσουμε και χρόνο και θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν δέχομαι το επιχείρημα που λέει ότι θα έχουμε επικαλύψεις και διπλές μετρήσεις και διπλή λογιστική. Πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο για το μεθάνιο και την αμμονία και να τα περιλάβουμε στην οδηγία. Και οποιαδήποτε μείωση των ρηπαντών αυτών είναι ευπρόσδεκτη και για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα αλλά και για την ποιότητα ε, του κλίματος γενικότερα. Τώρα, η φιλοδοξία μας νομίζω θα μπορούσε να είναι πιο αυξημένη. Αν δείτε τις τροπολογίες που ζητούν 67% στη σχέδια έκθεσης, εγώ θα ήμουν πιο φιλόδοξος, 75% θα έλεγα. Οικονομικά αυτό είναι πιο πρόσφορο. Και σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και σε σχέση με τις οικονομίες που θα κάναμε, ε, από 8,4 μέχρι 50 δις το, το χρόνο. Είναι σημαντικά το ωφέλη ε, για τα ε, συστήματα υγείας. Αφήστε δε που ε, μιλούμε και για 140.000 ζωές που θα σώζονται το χρόνο. Δεν είναι μόνο οικονομικό λοιπόν το όφελος. Για τους στόχους του 2020 Πρέπει να το συζητήσουμε και αυτός, γιατί υπάρχει και το πρωτόκολλο του Γκέτεμπορκ που ε, χωράει κάποια βελτίωση σε ορισμένε περιπτώσει. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη αυτή η προσπάθεια και από πλευρά σχεδιασμού 2020 ουσιαστικά είναι αύριο. Αλλά να μην το παραμελήσουμε και αυτό από τη συζήτηση. Και ένα τελευταίο θέμα. Παρόλη την κοινή μας προσπάθεια και το συνδυασμό δυνάμεων, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και ένα βασικό ρηπαντι που είναι ο υδράργυρος. Ορισμένοι ε, κλάδοι και τομείς εκπέμπουν υδράργυρο και δεν ξέρω γιατί έχει αυτό εξαιρεθεί. Έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στο νευρικό σύστημα, στο ανοσοποιητικό σύστημα, ακόμα και στο αναπαραγωγικό. Δεν θα πρέπει καθόλου να παραμελούμε τον υδράργυρο. Thank you very much. And now, Ms. Barter. Ευχαριστώ, η κυρία Μπίρτερ. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να πω πόσο ευτυχείς είμαστε που μπορούμε συλλογικά να συζητήσουμε την έκθεση αυτή ε, στην Επιτροπή σήμερα. Περιμέναμε πολύ και φαντάζομαι πως οι σκιώδες θα συμφωνούν ότι είμαστε ευτυχεί που επιτέλους μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα. Είναι ένα θέμα επί το οποίο η Κομισιόν εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και ξέρω πόσο χρόνο αφιέρωσε η Τζούλη και οι υπόλοιποι σκιώδει, αλλά και πολλοί έξω εκεί ε, ε, λομπίστε, ώστε να εξασφαλίσουν ότι δεν θα αποσυρθεί αυτή η έκθεση. Τώρα μπορούμε να αναπνεύσουμε πιο ήρεμα αφού έχει έρθει στην Επιτροπή μας η Επιτροπή. με δε που δεν μπορούμε να κάνουμε παρόμοιες συζητήσεις για την κυκλική οικονομία. Γιατί βούλιαξε το θέμα. Όλοι γνωρίζουμε τι αντίκτυπο έχει η κακή ποιότητα του αέρα στην ανθρώπινη παραγωγικότητα, στο περιβάλλον και η ποιότητα του αέρα ε, ε, ε, καλύπτει την πρωτοσέλιδα όχι μόνο εδώ αλλά και στην Κίνα, στην, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, σε ολόκληρη την Ευρώπη η ατμοσφαιρική ρήπανση προκαλεί 400.000 πρόωρους θανάτους. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει εκτιμηθεί ότι περίπου το 1 τρίτο της ατμοσφαιρικής ρήπανσης προέρχεται από την υπηρετική Ευρώπη. Η ατμοσφαιρική ρήπανση κοστίζει ζωές αλλά και χρήματα. Και γνωρίζουμε ότι σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει οι κυβερνήσεις να παίξουν το ρόλο τους στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Αν ήταν το πόσιμο νερό, που, ε, που, βγαίνει από τις βρύσες και ήταν τόσο μολυσμένο όσο ο αέρας, ε, τότε θα ενεργούσαμε μάλλον γρηγορότερα από ότι ε, τώρα, τόσα χρόνια που πήρε για να έρθει αυτή η έκθεση στην Επιτροπή μας. Συμφωνώ με την Τζούλη όσον αφορά την υποχρεωτική μείωση και τον συγκεκριμένο στόχο για το 2025. Αν τα αφήσουμε μέχρι το 2030 είναι πολύ σπάνιο, μάλλον πολύ απίθανο οι κυβερνήσεις ε, τοπικές, εθνικές και τα λοιπά να ασχοληθούν όπως πρέπει. Επίσης θα πρέπει να ζητήσουμε ενίσχυση του Euro 6, την πρόσφατη έκθεση δηλαδή από το Συμβούλιο για τη Μετασορές, γιατί οι εκπομπές ε, μονοξιδίου του ασώτου ε, εκτιμήθηκε ότι ήταν ε, έξι φορές μεγαλύτερες από ό,τι το επιτροπόμενο όριο. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Κομισιόν και η Κομισιόν θα πρέπει να επιπλήξει τα κράτη-μέλη που δεν συνεργάζονται στο Συμβούλιο. Για τους ρήπους. Θα ήθελα εδώ να έχουμε με περισσότερες φιλοδοξίες. Πρόσφατα στοιχεία από μελέτες αντικτύπου της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου δείχνουν ότι μπορούμε να μειώσουμε τους ρήπους γρηγορότερα και μέχρι το 2030 και με πιο οικονομικό τρόπο θα πρέπει αυτό να μας ε, δείξει, να μας οδηγήσει σε κλείσιμο του κενού κατά 75%. Ε, είναι ρεαλιστικό λοιπόν, θέλουμε να πάμε στις διαπραγματεύσεις με αυτά όλα και αυτοί που όλοι μας επιθυμούμε είναι καθαρός αέρας. Αν λοιπόν δεν προχωρήσουμε με φιλόδοξη εντολή στις διαπραγματεύσεις, ε, δεν θα μπορέσουμε να αντισταθούμε και να σταθούμε ε, στις θέσεις μας απέναντι στο Συμβούλιο. Τώρα, για τις δεσμευτικούς στόχους, για την αμμονία και το μεθάνιο. Ε, περιορίζονται μέχρι το 2030. Ορισμένε όμω χώρε, όπω η Ολλανδία έχουν τεράστια επιτυχία και έχουν μειώσει την αμμονία πάνω από 50% τι τελευταίε δεκαετίε. Ενώ άλλε χώρε είναι πολύ πίσω και το να το ζητήσουμε να κάνουν κάτι μόνο μέχρι το 2030 δεν είναι εφικτό. Επίσης, αναθεώρηση τη ΚΑΠ. Εγώ πιστεύω πως ε, αν δεν βάζουμε, βάλουμε εδώ στην νομοθεσία αυτά τα ζητήματα και η ΚΑΠ δεν τα αναθεωρήσει τα όρια, τότε χάσαμε το τρένο. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αναγνωρίσουμε την καλή δουλειά που έχουν κάνει ορισμένε χώρε και να στηρίξουμε άλλε χώρε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουν και εκείνε να ε, δουλέψουν. Επίσης, εξακολουθώ να ανησυχώ για τον ορισμό των μικρών ε, αγροκτημάτων και ποιος θα περιλαμβάνεται και ποιος όχι. Και τέλος, για την μεταφορά. Μπορώ να δω ε, τις μεταφορές. Ε, εντάξει, μπορεί να έχει νόημα να βγει από αυτή την ε, έκθεση, αλλά θα πρέπει να το εξετάσουμε, γιατί οι μεταφορές προκαλούν τεράστιους ρήπους. Αν θα το αναλάβουμε εμείς την πρωτοβουλία ή όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Πάντως, ε, ρηπαίνει και την ατμόσφαιρά μας. Αυτή η έκθεση νομίζω πως θα αυξήσει τις πράσινες θέσεις εργασίας. Η πράσινη οικονομία μπορεί όντως να καλύψει πολλές θέσεις και είναι καλό για τις επιχειρήσεις, είναι καλό για τις θέσεις απασχόλησης, είναι καλό για την ανθρώπινη υγεία και την ευημερία. Οπότε και πάλι να ευχαριστήσω την Τζούλη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 αν δεν ήταν τόσο πεισματάρα η Τζούλη, και το λέω με την καλή έννοια, δεν θα είχαμε την έκθεση αυτή σήμερα. Και, το, και εκείνη πίεσε, πίεσε με πείσμα και σταθερότητα, πήγε στην Επικομισιόν και εξασφάλισε ότι θα εξετάσει η έκθεση αυτή, ε, ότι θα εξεταστεί μάλλον αυτή η έκθεση Και γι' αυτό θέλω να την ευχαριστήσω που έχουμε σήμερα στην ημερησία μας διατάξει αυτή την έκθεση. Βέβαια η ποιότητα του αέρα θα πρέπει να είναι προτεραιότητά μας, αλλά και προτεραιότητα ολόκληρης της Ένωσης. Η ατμοσφαιρική ρήπανση δεν σέβεται τα σύνορα και έχει άμεση επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία τελευταία χρόνια είχαμε μια κάποια επιτυχία στην μείωση των εκπομπών, ιδιαίτερα από την βιομηχανία, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να αγωνιστούμε για ακόμα πιο καθαρή ατμόσφαιρα, να πιέσουμε ώστε όλοι να μπορέσουν και να υιοθετήσουν αυτούς τους νέους κανόνες. Θέλω να το τονίσω ότι οι συνθήκες στα κράτη-μέλη αλλάζουν με παρόμοιο βηματισμό και ρυθμό. Άρα λοιπόν δεν ζημιώνεται ε, κανείς περισσότερο από άλλους. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη. Ακόμα και η Γερμανία ή η Γαλλία δεν ανταποκρίνονται ούτε στις σημερινές προϊσχύουσες προδιαγραφές για, το, για τις εκπομπές. Θα πρέπει λοιπόν να συμφιλειωθούμε με το γεγονό ότι πρέπει να αναγκάσουμε κάποια, να πιέσουμε κάποια να κάνουν κάτι και για, σε άλλα ε, να ανεχτούμε ότι μπορούν τελικά να παρακάπτουν τις ε, υποχρεώσεις τους και να δημιουργούν εναλλακτικά μέτρα τα οποία δεν οδηγούν και σε πολλά σε σχέση με τα ε, καθαρή ατμόσφαιρα. Δεύτερον, τι θα μειωθεί και πόσο. Θείο, η οδηγία προτείνει ε, μείωση κάτω από το φυσικό όριο παραγωγής θείου. Για παράδειγμα, μόνο τα Ιταλικά ηφαίστεια το 2012 παρήγαγαν 2,5 εκατομμύρια τόνους θείου, ενώ ο ολόκληρος ενεργειακός τομέας ε, παρήγε 2 εκατομμύρια μόνο τόνους θείου. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε αν καταφέρουμε ρεαλιστικά, δηλαδή στην πραγματική ζωή, να τηρήσουμε αυτά τα όρια και τους στόχους. Ε, χαίρομαι για αυτό που είπατε για τις εκπομπές σκόνης, ιδιαίτερα τα σωματίδια ε, PM2,5 που είναι πολύ ε, επικίνδυνα για τον άνθρωπο και δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να τα εξαλείψουμε. Ένα άλλο θέμα που ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι είναι ο χρονισμός, δηλαδή οι ημερομηνίε και οι προθεσμίες. Ιδιαίτερα εδώ θα ήμουν εγώ υπέρ του 2030 ως ε, ε, στόχο. Το 2025 να είναι ένα ορόσημο ενδεικτικό και μόνο, αλλά όχι με δεσμευτικούς στόχους. Διότι ε, αυτό το θέμα συνδέεται πάρα πολύ με την τεχνολογική ανανέωση που χρειάζεται περισσότερο από πέντε χρόνια και πολλά κράτη-μέλη έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις και ακριβές και τεχνολογικά δεν θα είναι έτοιμα να φτάσουν στους στόχους μέχρι το 2025 από πλευράς υποδομών και μόνο. Επόμενο θέμα, η μείωση του διοξιδίου του άνθρακα και αντίστοιχη στόχη, ε, που είναι πάλι για το 2030. Κάτι που μου λείπει από την έκθεση αυτή και έχω κάπως απογοητευτεί είναι τι γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανανέωση της ε, μόνωσης στα σπίτια. Γιατί και αυτό θα βοηθήσει στη μείωση εκπομπής ρήπων. Πρέπει να μας απασχολήσει πιο λεπτομερώς και πιο σοβαρά. στους τριμερείς διαλόγους θα με ενδιαφέρει να ακούσουμε για αυτά τα θέματα, ιδιαίτερα από πλευρά Συμβουλίου, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που κάνουν προσπάθειες να φτάσουν σε αυτούς τους στόχους, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρουν έτσι ρεαλιστικά και αν θα προλάβουν στους χρόνους που εμείς ζητούμε να τα έχουν όλα αυτά υλοποιήσει. Επίσης, θα ήθελα η οδηγία αυτή να εναρμονιστεί με την οδηγία που μειώνει τις εκπομπές ρήπων στη βιομηχανία. Δεν ξέρω εάν αυτά που προτείνουμε είναι συμπληρωματικά ή αντιφατικά σε κάποια σημεία και θα ήθελα να με διαφωτίσετε σχετικά. Ένα τελευταίο θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί οι ρήποι που θέλουμε να μειώσουμε. Ας πούμε, η θέρμανση τοπική σε κάποιες περιφέρειες, σύμφωνα με μελέτες, ευθύνεται ε, μέχρι και για το 1 τρίτο των ε, ρήπων σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση δηλαδή. Εάν θέλουμε ρεαλιστικά να μειώσουμε τις εκπομπές ε, των μεταφορών, θα πρέπει να επικεντρωθούμε όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά και στην θέρμανση κατά τόπους, γιατί ε, είναι ο τρίτος ε, ρήπος και πηγή ρήπασης ε, κατά σειρά. Σε ό,τι αφορά τώρα την αυτιλία, τις θαλάσσιες μεταφορές και τα αντίστοιχα όρια ή την αύξηση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στις πόλεις και άλλα, Υπάρχουν διάφορες προτάσεις για περιφέρειες χαμηλής ρήπασης. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία προτάσεις, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ρεαλιστικά αν σκεφτούμε πώς είναι σήμερα οι πόλη μας. Και ας κοιτάξουμε περισσότερο τη θέρμανση και τους μικρούς εκπομ... Ε, τις μικρές εκπομπές ρήπο, ε, για να προλάβουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ όλους και όλους οι και την εισηγήτρια. και θα πρέπει με λογική να προχωρήσουμε και τελικά πιστεύω ότι θα βρούμε μια κοινή λύση και μια λογική λύση. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now Mr. Pedicini. Ο κύριος Πεντιτσίνη τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον συνάδελφο Γκέρλινγκ για την δουλειά που έκανε ως εισηγήτρια. Κυρίως αν σκεφτούμε την καθυστέρηση και την αβεβαιότητα που είχαμε για κάποιο διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η οδηγία αυτή, αν θέλουμε να στραφούμε προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, για να προστατεύσουμε και την υγεία και το περιβάλλον. Το πακέτο αυτό όμως θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη να περάσουν σε άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας από ό,τι τα στερεά καύσιμα. Ένα σύστημα ελέγχου λοιπόν χρειάζεται, ένα μόνιμο σύστημα που θα διασφαλίζουν και ανεξάρτητοι και αναγνωρισμένοι οργανισμοί οι, οποία, οι οποίοι σε, ε, σε πραγματικό χρόνο θα δίνουν πληροφορίες και τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν λοιπόν στην έκθεση αυτή πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία κατά τη γνώμη μας. Το θέμα του δεσμευτικού στόχου του 2025 συμφωνούμε, συμφωνούμε και για τις δοκιμές όσον αφορά τα οχήματα που μπαίνουν στο εμπόριο. Συμφωνούμε επίσης και για τις πιο πρόσφατες κατηγορίες, για τα αποτελέσματα. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Συμφωνούμε και για το θέμα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη όπως και για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2020, αν και για μας χρειάζονται ειδικέ δράσεις για την περίοδο 21 μέχρι 27. Εκεί που διστάζουμε περισσότερο είναι για την αμμονία. Θα αξιολογήσουμε πάντως πιο προσεκτικά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Φλόρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά εγώθηκαν και πολλά σωστά και επενετικά και σωστά την ε, επενούν την εισηγήτρια. Συμφωνώ και εγώ με μεγάλη χαρά διοργανικά. Η ρήπανση ε, ε, είναι διεθνής. Δεν γνωρίζει σύνορα και σε δική μου χώρα, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Και εμεί δεν ε, έχουμε πολύ καλές επιδόσεις στη Γερμανία, ιδιαίτερα για την αμμονία. Αλλά βλέπουμε πολλά τα κράτη-μέλη ε, είναι αυτά που δεν έχουν καταφέρει τους στόχους. Γιατί? Ε, όχι μόνο στην αμμονία που είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, αλλά και αλλού. Γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι σωστές οι νομικές προϋποθέσεις και οι συνθήκες που δημιουργούν και το πλαίσιο γιατί επιτρέπουμε τα παραθυράκια και σε διαφόρους να ελίσσονται και να διαφεύγουν. Και έρχομαι αμέσω στο θέμα του υποχρεωτικού ημί. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το 2025 είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Ακόμα και αν με κυνηγήσουν οι αγρότες μου. Αλλά αν αφήσουμε τους στόχους για το 2025 προαιρετικούς θα προσπαθήσουν όλοι μέχρι το 2029 να αναβάλουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν και το 2030 θα αρχίσουν να τρέχουν και θα λένε αμάν δεν προλαβαίνουμε. Και αν δεν με πιστεύετε εμένα, ρωτήστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ξαναρωτήστε με εμένα. Έχει επανειληφθεί αυτό πολλές φορές σε διάφορες περιπτώσεις δείξαμε αυτή την ανοχή την οποία εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι προς μια κατεύθυνση που δεν μας άρεσε. Οπότε Εντάξει, να είναι δεσμευτική με μέτρο, δεν μπορεί να πάρουμε μια βαριοπούλα και να αρχίζουμε δεξιά και αριστερά να ε, χτυπάμε. Και ε, σταματάω λοιπόν, θα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια κοινή προσέγγιση. Τα τελευταία δέκα χρόνια είχαμε επικεντρωθεί στο ε, διοξίδιο του άνθρακα και παρενοχλήσαμε μέχρι ε, εκεί που δεν πάει την βιομηχανία ενώ ε, τους αγρότες και τα νοικοκυριά τα βλέπουμε μεγαλύτερη επίοικια. Ε, θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Και δεν μπορούν ε, ορισμένοι να έχουν ιδιαίτερα ε, χαλαρή προσέγγιση και κάποιοι άλλοι να είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Ε, Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική αναφορά, θα ήθελα να πω στην κυρία Γκέρλινγκ ότι εγώ δεν είμαι κατά ανάγκη κατά. Στη χώρα σας χρειάζεται μία μόνο, στη δική μου χώρα χρειάζεται 15, συν το Βερολίνο μία 16, κεντρική κυβέρνηση, για να στείλουμε ε, στις Βρυξέλλες. Και εγώ ρωτώ, έτσι με κάθε φιλικό πνεύμα, για ποιο λόγο να υπάρχει υποχρεωτική αναφορά. Επανειλημμένα έχουμε ζητήσει εμείς, αμέτρητες υποχρεωτικές αναφορές και εγώ ο ίδιος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συμπεράσματα εξάγει μετά και τι συνέχεια δίνει, τι τα κάνει όλα αυτά που τις στέλνουμε υποχρεωτικά. Όταν κάνω εγώ ένα νόμο ας πούμε. Τελικά τι αποτέλεσμα έχει, θέλω να δω είναι η τόπο όλος αυτός ο κόπος. Τι όλοι να ανοίξουν τα σχήρα τους και να έχουν τη δικαιολογία τους. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολη αυτή η συζήτηση. Αύριο το πρωί αρχίζει από την πολιτική μου ομάδα αυτή η δυσκολία. Αλλά μόνο από κοινού θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και εδώ όλους τους κλάδους της οικονομίας. Δεν θα πρέπει να εξακολουθούμε να είμαστε κατακαιρματισμένοι, γιατί το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να τσακωνόμαστε μεταξύ μας και θα καταλήξουμε σε σούπερ φιλελεύθερες αποφάσει, ε, ευνοϊκές υποτίθεται για όλα τα κράτη-μέλη και μετά τα μισά από τα κράτη δεν θα κάνουν τα μαθήματά τους. Ας είμαστε λίγο πιο μέτριο παθή στις τιμές να τις στηρούμε και όμως. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βίτεμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια εισηγητή από την Επιτροπή Γεωργία. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πολύ ευχάριστη και καλή συνεργασία μέχρι τώρα μαζί τη. Από τη Επιτροπή Γεωργία, λοιπόν, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο σημεία. Το ένα είναι η αμμονία βέβαια και το άλλο είναι ε, το διάμεσο στάδιο. Και το μεθάνιο, συγγνώμη, και το μεθάνιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουμε διάκριση ανάμεσα τους ε, ρηπαντές, τις δεπογόνες ουσίες και τα αέρια του θερμοκηπίου. Έχουμε από τη μια μεριά το ETS και από την άλλη μεριά έχουμε το MCP και την οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών που προπαλεί να προσπαθούμε μάλλον να ε, συμπεριλάβουμε και άλλα αέρια του θερμοκηπίου σκηνοβούλου, αλλά τελικά είπαμε όχι. Και τώρα ε, γίνεται το αντίστροφο, δηλαδή ε, συμπεριλαμβάνουν το μεθάνιο. Φοβούμε λοιπόν ότι θα γίνει διπλός κανονισμός εδώ και αυτό θα οδηγήσει σε έλλειψη ευελιξίας. Για να δώσω ένα παράδειγμα στον τομέα τον γεωργικό τα, οι εκμεταλλεύσεις ε, γεωργικές μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν όσον αφορά την, κατακράτηση των αερίων του θερμοκηπίου όπως ας πούμε το διοξίδιο του άνθρακα. Πρόκειται για, φυτε, για χορτολιβαδικές εκτάσεις που είναι σημαντική σημαντικές λεκάνες απορρόφησης διοξιδίου του άνθρακα. Ε, εμείς δηλαδή στην ουσία τι κάνουμε, θα τους τιμωρήσουμε επειδή εκπέμπουν μεθάνιο αλλά δεν θα τους ανταμείψουμε επειδή συλλέγουν ε, και κατακρατούν άλλα αέρια του θερμοκηπίου. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ευελιξία ώστε οι γεωργοί να μπορούν να συμβάλλουν έτσι στην ε, απάλυνση των επιπτώσεων και των κλιματικών αλλαγών. Ένα άλλο θέμα είναι ε, το θέμα των βοσκοτόπων. Εάν θέλουμε να μειωθεί το μεθάνιο, ιδιαίτερα στο τομέα των γαλακτοκομικών, θα πρέπει να αφήνει τα ζώα σου έξω ε, ολόκληρο το χρόνο και το να βρίσκεις χορτολιβαδικές εκτάσεις είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και είναι δύσκολη η επίτευξη τη μείωση του μεθανίου. Για την αμμονία, όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι κρατημέλοι έχουν επενδύσει ήδη πολλά στην μείωση της τη αμμονία, αλλά όχι. Ε, Ορισμένοι λοιπόν, έχουν κάνει λοιπόν τεράστιες προσπάθειες. Εγώ στη δική μου έκθεση θέλω να καταστήσω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε, όπως είπε ο κύριος Φλόρεντς, σε ένα ισότιμο πεδίο. Ε, δηλαδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβάλουν τις ίδιες ε, ε, προσπάθειες σε σχέση με την αμμονία όλα και αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στην πρόταση της Επιτροπής. Επίσης προσβλέπω σε συζητήσεις ε, που θα γίνουν εδώ και να... Έχω και άλλες παρατηρήσεις για την ΚΑΠ, αλλά ε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι να συζητήσουμε εις βάθος την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, η κυρία Σχράερ Πίρικ. Συγχαρητήρια στην κυρία Γκέρλινγκ είναι μια έκθεση που με ενδιαφέρει πολύ και όχι μόνο εμένα, αλλά παρακολουθούν και πολύ στην Ολλανδία την έκθεσή σας. Εγώ είμαι σχιώδης εισηγήτρια, ε, όπως και ο κύριος Χαϊτεμα, συμφωνώ με αυτά που είπε. Για την αμμονία θέλω να μιλήσω κι εγώ. 30% μείωση, αλλά στην ε, Ολλανδία είχαμε 66% αύξηση. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε σε μηδενική βάση από το 2005. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και πολλές οικονομικές επιβαρύνσεις ήταν αυτές για τους αγρότες ε, και προηγούμενες και σημερινές ε, προσπάθειες για τη μείωση της αμμονίας θα πρέπει να αναγνωριστεί όπως το αξίζει για να υπάρχει τότε μόνο ένα ε, ίσο πεδίο. Αλλιώς δεν πρόκειται να σας ακολουθήσουν οι ε, Και το θέμα της ευημερία των ζώων είναι πολύ σημαντικό και μπορούμε να επιτύχουμε πολλά. Αλλά όταν πρόκειται για δεσμεύσεις, για την αμμονία σε συνδυασμό με το μεθάνιο στην πρόταση, ε, τότε αυτό δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες. Το είπε μόλις ο κύριος Χάιτεμα και συμφωνώ απολύτως. Ε, συγκράτηση διοξιδίου του άνθρακα, αλλά ήθελα να μιλήσω και για κάτι άλλο. Ε, οι συνάδελφοι του Σοσιαλιστικού Κόμματος τι λέτε, πηγαίνετε σε όλη την Ευρώπη και δεν βλέπετε πουθενά αγελάδα ε, σε ένα λιβάδι. Ούτε στην Ολλανδία ούτε στην Αυστρία να εξαφανιστούν από παντού οι αγελάδε και δεν υπάρχει ένα τοπίο με βοσκοτόπους. Το είπε και ο κύριος Τίμερ μας εδώ, ο α, αντιπρόεδρος. Η, η μείωση δεν μπορεί να είναι μόνο ένα αποτέλεσμα υποχρεωτικής νομοθεσίας, θα πρέπει να το δούμε και από άλλο. θα πρέπει να είναι πιο αναλογικές και σωστές οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε διάφορους κλάδους της οικονομίας ε, και στην αναψυχή και στις μεταφορές και στη βιομηχανία με αντίστοιχο τρόπο να συνεισφέρουν όλοι στη μείωση της ε, ε, ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, ιδιαίτερες επιβαρύσεις στους γεωργούς. Είναι άδικο αυτό γιατί έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες τις τελευταίες δεκαετίες. Έχω κάνει τροπολογίες και έχω ζητήσει και από την εισηγήτρια να βρεθούν ε, κονδύλια για τη γεωργία για αγρότες που κάνουν πολύ σοβαρές προσπάθειες εδώ και χρόνια σε αυτό το δομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Όχι. Α, παρακαλώ. Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης είναι συνδεδεμένο άμεσα και με την οικονομική κρίση ο τομέα τη θέρμανση, που είναι μαζί με τα καυσαέρια των αυτοκινήτων μια μεγάλη πηγή ρήπανση, πρέπει να εξεταστεί. Λόγω τη οικονομική κρίση και τη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο στην Ελλάδα, οι πολίτε, προκειμένου να ζεσταθούν, στράφηκαν σε άλλε πηγέ, όπω τι ξυλόσομπε και στα τζάκια. Όμω, επειδή και τα καυσόξυλα ήταν ακριβά ή δεν είχαν χρήματα για να αγοράσουν, έκαιγαν τους προηγούμενους χειμώνες ό,τι έβρισκαν. Παλιά έπιπλα, πόρτες, παράθυρα. Οι εθάλοι και τα μικροσωματίδια έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια του συναγερμού. Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις, την κυριολεξία. Όμως, από την κάψη αυτών των υλικών, τα οποία είχαν πάνω βερνίκι και χρώματα, ο αέρας δηλητηριάζονταν στην κυριολεξία από χημικές ενώσεις άκρω επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Ήδη τα κρούσματα με ασθένειες που αφορούσαν το αναπνευστικό είχαν εκατοντοπλασιαστεί. Το φυσικό αέριο που είναι σχετικά πιο καθαρή μορφή καυσίμου στην Ελλάδα δεν υπάρχει δίκτυο που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει όλες τις κατοικίες. Έτσι η κατανάλωση φυσικού αερίου είναι μικρή και η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμα γιατί δεν καταναλώνει ετησίως το αέριο που έχει συμφωνήσει. Η οικονομική κρίση λοιπόν συμβάλλει και στη ρήπανση της ατμόσφαιρας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Αν δεν υπάρχει κανείς άλλος που θέλει το λόγο, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Ποιον έχουμε από την Επιτροπή? Την κυρία Βένινγκ. Παρακαλώ, για να απαντήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Θέλω Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Γκέρλινγκ, την εισηγήτριά σας, για μια πολύ πλήρη έκθεση που παρουσιάζει και καλά ισορροπημένη θα έλεγα, η οποία σε μεγάλο βαθμό στηρίζει την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θέλω να επαναλάβω, Πρόεδρε, εδώ, ότι μετά τα όσα έγιναν την τελευταία εβδομάδα σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θα έλεγα ότι σήμερα είναι ακόμα πιο σημαντικό το ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές και αυτό με αποτελεσματικό τρόπο. Οι τελευταίες εβδομάδες, η ρήπανση που διαπιστώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν κάτι μεμονωμένο, το συναντάμε όλο και πιο συχνά. Και αυτά είναι ακριβώς που μας πείθουν για το ότι πρέπει γρήγορα να προχωρήσουμε στην μείωση των ρηπογόνων ουσιών και να πετύχουμε τους στόχους μας. Έχουμε λοιπόν τη φιλοδοξία και εμείς να μειώσουμε την ατμοσφαιρική ρήπανση, να μειώσουμε τις επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων πάνω από 50%. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε γι' αυτό και θέλουμε να το κάνουμε με όσο γίνεται μικρότερο κόστος, πετυχαίνοντας όμως τους στόχους μας. Έτσι κι αλλιώς η ζημιά μας κοστίζει 10 φορές παραπάνω από όσο μας κοστίζει η αντιμετώπιση του φαινομένου. Επιτρέψτε μου τώρα να σας δώσω κάποια σχόλια, όχι τόσο επεξηγήσεις, για τα πιο σημαντικά ζητήματα κατά τη γνώμη μας που θέτει η συγγήτρια αλλά και άλλα μέλη της Επιτροπής σας. Αρχίζω με το θέμα της αμμονίας και των υποχώνων ουσιών περιλαμβάνονται στην πρόταση αυτή. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι οι στόχοι για τις ουσίες αυτές παραμένουν στην πρόταση. Και θέλουμε να απαντήσουμε στις ανησυχίες που εκφράσατε. Όταν είχαμε την ε, ανησυχία για ένα διπλό κανονισμό ε, ενέργεια και κλίμα, δεν ισχύει. Η πρότασή μας έγινε σε απόλυτο συντονισμό με το θέμα της ενέργειας ε, και του κλιματικού πακέτου. Είναι οι ίδιες δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε και εκεί. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι οι επιλογές αυτές είναι χωρίς κόστος. Λέγαμε ότι 4 δισεκατομμύρια μπορούν να κερδίσουν οι αγρότες από την μείωση των εκπομπών και είναι κάτι που δεν ε, εμποδίζει καθόλου τη δικιά τους την ευελιξία ή τη γενικότερη ευελιξία του πακέτου. Από πλευράς ευημερία που και αυτό αναφέρθηκε και έχει να κάνει και με την αμμονία, θα πρέπει να βρούμε μια καλή ισορροπία, όπως βέβαια πρέπει να κάνουμε πάντα. Πάντως δεν θα πρέπει να βάλουμε το ένα θέμα σε ανταγωνισμό με το άλλο, αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Δεν είναι το θέμα ε, της προστασίας ε, των ζώων, για παράδειγμα, από τη μία και το άλλο, το θέμα της μείωσης των ρηπογόνων ουσιών. Αμμονία τώρα. Ε, Προέρχεται σε 90% πολλές φορές από την γεωργία. Πολλοί από εσά αναφερθήκαν στις προσπάθειες που έχουν κάνει και άλλες κοινωνικές ομάδες, η ίδιομηχανία, τα νοικοκυριά. Θέλω να υπενθυμίσω ότι προς το παρόν δυστυχώς η μείωση στην Αμονιάρα και στη Γεωργία ήταν πολύ χαμηλή. Η πρόοδος δηλαδή που έγινε για τη μείωση των εκπομπών αμμονίας ήταν ελάχιστη. Όταν έχουμε 80% για το διοξίδιο του άνθρακα, ας πούμε, έχουμε 20% μόνο για την αμμονία. Και αν δούμε και το κόστος που πήγε στην μείωση των βιομηχανικών εκπομπών και των γεωργικών εκπομπών, πάλι έχουμε ποσοστά, το οποίο δείχνουν ότι είναι 47% στη μία περίπτωση, 2% στην άλλη. Για να υπάρχει λοιπόν η ίδια αντιμετώπιση όλων των τομέων, πρέπει να κάνουμε κάτι και στον τομέα της γεωργίας. Καταλαβαίνουμε ότι οι γεωργοί εκφράζουν ανησυχίες. Πιστεύουμε όμως ότι με την τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, και εδώ μάλιστα και αρκετό καιρό ήδη, μπορούμε κάλλιστα να πετύχουμε τους στόχους που προτείνουμε. Και επειδή φαίνεται ότι αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τις χώρες μέλη, αυτό δεν είναι αλήθεια. Αν δούμε από το 1990 μέχρι το 2030, ε, θα δούμε. Όντως, οι χώρες που πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια ε, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα, αλλά είναι σημαντικό να σας δώσω την προοπτική χρονικά, δηλαδή, για την οποία μιλάμε. για τους δεικτικούς ε, δείκτες που συζητάμε για το 2025. Και ακούσαμε εδώ ότι πολλοί από εσά θέλουν να είναι υποχρεωτικοί αυτοί, εκτός από την αμμονία. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τα επιχειρήματα που ακούστηκαν και εδώ σήμερα. Και πάλι όμως πρέπει να σκεφτούμε το 2030 και τους στόχους που τότε θα πρέπει να έχουμε πετύχει. Κάποιοι από εσά είπαν ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον επενδυτικό κύκλο. Ναι, συμφωνούμε και αυτό προτείνουμε. Να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που είπε ο κύριος Φλόρεντς δεν θα γίνει. Ότι δηλαδή οι χώρες μέλη δεν θα περιμένουν την τελευταία στιγμή για να προσαρμοστούν. Γι' αυτό θέλουμε και ένα ενδιάμεσο στάδιο. Θέλουμε σιγά σιγά να γίνεται ο έλεγχος, ώστε όσοι δεν κάνουν αρκετά να εντοπιστούν. Βάζοντας για το 2025 δεσμευτικούς στόχους θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να μην βρεθούμε σε αδιέξοδο και να προχωρήσει ο παιδιτικός κύκλος κανονικά. Θέλω να αναφερθώ και στην ευελιξία στις εκπομπές των θαλασσίων μεταφορών που ξέρετε ότι είναι κάτι που έχει πάρει μεγαλύτερο μέγεθος γιατί οι χερσαίες μεταφορές πάντα κυριαρχούσαν στις συζητήσεις για την μείωση των εκπομπών τις τελευταίες δεκαετίες. Οπότε στον υπολογισμό των εκπομπών των θαλασσίων μεταφορών δεν δίναμε εξίσου σημασία παρόλο που και αυτές οι, μεταφορε... εκπομπές μεταφέρονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρόλο που μπορεί να δημιουργούνται στη Βόρεια Θάλασσα, για παράδειγμα, οι επιπτώσεις της ρήπανσης αυτής γίνονται, γίνονται σε πολύ περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι χώρες μέλη λοιπόν θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και αυτό το στοιχείο τους στόχους. Δεν λέω εδώ ότι πρέπει να βάλουμε σε αντιπαράθεση τις χώρες που έχουν που δεν έχουν θάλασσα. Αλλά είναι μια πτυχή που σίγουρα πρέπει να ληφθεί υπόψη και θέλουμε και εμείς να τη διατηρήσουμε. Κάποια άλλα ζητήματα τώρα. Στηρίζουμε απόλυτα ότι το ότι πρέπει να υπάρχει οικονομική στήριξη για τους στόχους αυτούς. Υπάρχει και, στο, υπάρχουν και στα προγράμματα. Η μεταρρύθμιση της κοινή συλλογικής πολιτικής ε, το προβλέπει για δραστηριότητες των χωρών μελών που μπορούν να στηριχθούν οικονομικά. Συχνά βέβαια βλέπουμε ότι οι χώρες μέλη δεν το γνωρίζουν. Συνεπώς πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση για τα ποσά αυτά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές οι χώρες υπάρχουν. Το θέμα είναι οι χώρες μέλη να τα ζητήσουν για να τα χρησιμοποιήσουν. Όσον αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση και τη συμμετοχή, ναι, και αυτά είναι θέματα που είναι και για μας πολύ σημαντικά. Θα τα στηρίξουμε. Ένα άλλο στοιχείο, και νομίζω ότι με αυτό θα ολοκληρώσω, το πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τις δοκιμές, με τις αξιολογήσεις που γίνονται. Εμείς πάντα λέγαμε ότι θα το κάνουμε. Το κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις ανησυχίες των χωρών μελών, αλλά τους έχουμε πει, όπως το λέμε και σε εσά εδώ τώρα, ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος γρήγορα. Πρέπει για το πρώτο στάδιο ε, της αναθεώρησης ε, του κύκλου πρέπει να έχει εγκριθεί αυτό ώστε το 2017 να μπορέσει να εφαρμοστεί πλήρως η αναθεώρηση και να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο. Συνεπώς η στήριξή σας εδώ είναι πολύ σημαντική. Πρόεδρε, αυτά, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε έτσι να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για το σημείο αυτό, δίνοντας το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Κέρλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους σας. Φάνηκε από τη συζήτηση ε, ότι ε, τα σημεία που ανέφερα στην αρχή ως επίμαχα είναι εκείνα που χρειάζονται περισσότερη συζήτηση, ιδιαίτερα για την αμμονία. Καλό είναι όμως να ακούμε ότι το έχουμε εντοπίσει ως πρόβλημα και θα πρέπει να το συζητήσουμε και μάλιστα σε πολλές λεπτομέρειες για το πώς θα προχωρήσουμε. Είναι κρίμα και απογοητευτικό που δεν ακούσαμε τους πρασίνους. Διότι από τις συζητήσεις που είχα Έχανε κάποια θέματα να θέσουν ως προς την ε, φιλοδοξία. Το άφησαν στον κύριο Ντόνσον, το, καλά το χειρίστηκε, αλλά ε, μέχρι ενός βαθμού είναι τακτική και ακόμα πιο πέρα είναι στρατηγική. Ελπίζω οι σκιώδεις ηγητές θα συνεχίσουμε να συζητούμε αυτά τα θέματα για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Ε, θέλω να πω κάτι που ίσως έπρεπε να το είχα πει στην αρχή και είναι γενικότερο. Είναι μια κλασική περίπτωση νομοθεσίας όπου μέσο και μακροπρόθεσμα ε, είναι αμοιβαίως επωφελής. Δηλαδή μπορούμε να βελτιώσουμε και την υγεία και θα, θα μας κοστίσει θεωρητικά και τίποτα αν δούμε τα στοιχεία και τους αριθμούς. Αλλά είναι και μια χαρακτηριστική κλασική περίπτωση όπου το κόστος πέφτει σε ένα κλάδο της οικονομίας ενώ το όφελος αλλού χωρίς να φαίνεται πάντα. Και αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα, το πώς το διαβιβάζει στην κοινωνία. Ε, μπορεί να είναι το κόστος μηδενικό ή ακόμα και ωφέλεια, αλλά εκείνος που επομίζεται το κόστος δεν συμφωνεί πάρα πολύ, γιατί δεν είναι αυτός που θα έχει το όφελος τελικά ή θα είναι γενικότερο προς όφελος της κοινωνίας. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, όπως είπαμε, και γι' αυτό χαίρομαι πολύ που με υποστηρίζετε για να βρούμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε μέσω της διαδικασίας και τελικά να καταλήξουμε με τη σωστή λύση. Σας ευχαριστώ όλους και περιμένω με χαρά την επόμενη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Thank you to you. I have to... Εγώ σας ευχαριστώ. Πρέπει να θυμίσω εδώ το χρονοδιάγραμμα για το κείμενο αυτό. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 21 Απριλίου. Οι ε, τροπολογίες ε, θα συζητηθούν 16 και 17 Ιουνίου ε, στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε στην τελευταία συνεδρίαση του Ιουλίου μας στις 15 του μηνός. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση. Ε, η συνεδρίαση της Επιτροπής στις 5 ακολουθεί η συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ.